Um, they're going coming the Λοιπόν, περνάμε τώρα στα περίπλοκα. Ας προσπαθήσουμε να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Καταρχάς, να κάνουμε μία δοκιμαστική ψήφο, παρακαλώ, πρώτα. Λοιπόν, δοκιμαστική ψήφος, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. 39 κάρτες έχουν μπει στη θήκη, 37 έχουν πιεστεί, 38 έχουν πιεστεί. Ο Ζων Πολ ψάχνει τη δική του. Θα ήθελα να πω στους φιλελεύθερους ότι έχουμε ένα παραπάνω, ψηφίζω και εγώ, οπότε κάποιος από την Άλντ ίσως θα πρέπει να βγάλει την κάρτα του. ένας από τους αναπληρωτές των φιλελευθέρων δεν θα πρέπει να ψηφίσει. Λυπάμαι γι' αυτό. Λοιπόν, η πρώτη ψηφοφορία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 Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε για το FTT παρακαλώ, τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Λοιπόν, πρώτη ψήφος για την έκθεση της κυρίας Ποδηματά τροπολογίες 26 και 27 από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 28 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 1 με 4 υπέρ κατά αποχές δεκτό A, ε, α κεφαλαίο, υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Β κεφαλαίο, υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Σ αγγλικό, υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά αποχές δεκτό τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό στο F το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό στο G αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το I αγγλικό υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τροπολογία 9 υπέρ. Η 9 για μια στιγμή λέει η πρόεδρος, διακόπτη η πρόεδρος. Έχει καταπέσει η 9, συγγνώμη. Το πρωτότυπο λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Κάπα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα το αρχικό κείμενο στο μη υπέρ κατά αποχές δεκτό. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αρχικό κείμενο στο νη υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Όμικρον, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Οι επόμενες ε, τρεις έχουν καταπέσει. Επειδή έγινε δεκτή η 11, έχει καταπέσει και η 23 και η 24. Λοιπόν, 25 με προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια. Διαφωνεί κάποιος με την προφορική, όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 25 με την προφορική, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα ψηφίζουμε το τροπολογημένο κείμενο συνολικά, ηλεκτρονική ψήφος παρακαλώ. Δύο μπορούν να ψηφίσουν ακόμα πέρα της ψηφοφορίας. Λοιπόν βρήκαν όλη την κάρτα τους. 32 υπέρ, μία αποχή και 6 κατά. Ευχαριστώ πολύ την εισηγητρία.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 στην έκθεση φυσκάλη του Στόλογιαν. Καταρχάς, προϋπολογισμός 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προϋπολογισμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 33. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 με προφορική τροπολογία. Συμφωνείτε για την προφορική ε, τροπολογία. Λοιπόν, 41 ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική C είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11. Α, όχι, έχει καταπέσει 11. 45 έχει καταπέσει επίσης. Προϋπολογισμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική διαγλικό ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 έχει αποσυρθεί 13 προϋπολογισμός υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 εισηγητής υπέρ κατά αποχές δεκτή. 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική D, D υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ, έχει αποσυρθεί μάλλον η 62-63 με προφορική τροπολογία. Συμφωνείτε να κατατεθεί με προφορική τροπολογία. Καλώς ψηφίζουμε 63 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Προϋπολογισμός 14 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Προϋπολογισμός 15 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ή αγγλικό υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 με προφορική τροπολογία συμφωνείτε με την προφορική όχι 67 λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές δεκτή Η 48 έχει καταπέσει γιατί καλύπτεται από την προφορική τροπολογία. Προπολογισμό 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προπολογισμό 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προπολογισμό 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική F αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική G αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική αγγλικά H υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Α, όχι, συγγνώμη, έχει αποσυρθεί 26. Συμβιβαστική I αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική J αγγλική υπέρ κατά αποχές δεκτή Προϋπολογισμός 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η ηλεκτρονική ψήφος τώρα επί του συνόλου του τροπολογημένου κειμένου. Ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 40 υπέρ κανείς κατά μία αποχή. Τώρα ηλεκτρονική ψήφος επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Ψηφίζουμε. vote. Press your buttons again. Four more of you. Three. Λάτε. Τέσσερις παραπάνω. Δύο παραπάνω. Ένας παραπάνω. Κάποιος περισσεύει ή κάποιος δεν ψηφίζει. Πέρα της ψηφοφορίας. Τελείωσε. 40 υπέρ, καμία ψήφος ε, κατά, μία αποχή. Ωραία, μπορούμε να χειροκροτήσουμε. Τώρα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον συγητή. Ο εισηγητής μας ζήτησε να λάβει εντολή για τυχόν συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Θέλετε να πείτε δύο λόγια από αυτού. Όχι λέει ο κύριος Τόλογιαν. Απλώς θα ήθελα να ζητήσω, α, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες και είμαι ε, πολύ ευγνώμων για τη συνεργασία που είχαμε. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ πρόθεσή μας είναι να αρχίσουμε τις διαβουλεύσεις για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να συμφωνήσουμε στην πρώτη ανάγνωση σύμφωνα με την τακτική διαδικασία και η, διαβουλευτική, ομάδα διαβούλευσης θα αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο που είναι και εισηγητής. Ε, τον εισηγητή λοιπόν, τον σκιώδη εισηγητή και η εντολή θα ε, δοθεί για να ψηφιστεί σήμερα στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Τώρα αν είναι να τις προβάλλετε, αλλιώς θεωρούμε ότι έχει ότι ούτως θα προχωρήσουμε. Χωρίς ψηφοφορία. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, άρα συμφωνούμε όλοι σιωπηλώς. Να αρχίσουν οι διαβουλεύσεις. Δεν πιστεύω να αρχίσει ο τριμής διάλογος μέχρι το Φεβρουάριο λόγω του Συμβουλίου που δεν έχει ακόμα προχωρήσει. Πολύ ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο. we're now moving on to the, um, uh... Προχωρούμε στο πακέτο SSM και αρχίζουμε με την έκθεση Tyson, μετά προχωρούμε στην έκθεση Giggold. Δεν ξέρω αν ο Ζανπόλ θέλει να πει κάτι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να εκφράσουμε την άποψή μας για δύο πάρα πολύ σημαντικά έγγραφα. Βέβαια δεν έχουν την ίδια νομική, το ίδιο νομικό καθεστώς, δεν διέπει και τα δύο έγγραφα. Και από πλευράς Συμβουλίου υπάρχει μια κάποια σύγχυση Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας, ζητώ την αναβολή της ψηφοφορίας και των δύο εκθέσεων για τεχνικούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Πρώτον, πλέουμε στην ομίχλη σε ένα σύστημα το οποίο δεν έχει καθοριστεί ακόμα από τα κράτη-μέλη και ανάμεσά τους υπάρχουν σημαντικές διαφορές και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο τεχνικό και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το Κοινοβούλιο να ξεκαθαρίσει λίγο την ατμόσφαιρα. Και κυρίως την επόμενη εβδομάδα υπάρχει το ΕΚΟΦΗΝ το οποίο θα συνεισφέρει νέα στοιχεία στη συζήτηση και γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερος χρήσιμο αναζητώντας μια σωστή μορφή εργασίας και συνοχής της διαδικασίας να αναβάλουμε για λίγες εβδομάδες την ψηφοφορία των δύο αυτών εγγράφων. Εξ αρχής είχαμε δεχθεί να ακολουθήσουμε ε, θα έλεγα τη διαδικασία με υψηλή ταχύτητα γιατί αυτές ήταν οι προοπτικές μας. Είχαν πει ότι θα ήταν έτοιμα τα κείμενα την 1η Ιανουαρίου του 2013. Είναι προφανές ότι μια τέτοια προθεσμία δεν θα γίνει σεβαστή κατά από τις παρούσες συνθήκες λοιπόν. Θα ήταν χρήσιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην προτρέξει του Συμβουλίου και να μπορέσει το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να ελέγχει την κατάσταση και γι' αυτό ζητώ την αναβολή της ψηφοφορίας των δύο αυτών εκθέσεων υπογραμμίζοντας την εξαιρετική εργασία των δύο εισήγητων για να καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες στην παρούσα φάση την χάνουν πλειοψηφιών, στήριξη από πλειοψηφίες. Αλλά δυστυχώς όπως έχουν τα πράγματα ζητώ την αναβολή της ψηφοφορίας. Um, Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Τη βιασύνη την οποία αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε ε, λόγω πιέσεων. Τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει να ψηφίσουμε αμέσως, αν θέλετε, την αναβολή της ψηφοφορίας ή όχι των δύο αυτών ε, θεμάτων. Εάν ψηφίσετε ναι, τότε ε, σημαίνει ότι θα αναβάλουμε. Εάν ψηφίσετε όχι, σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε με την ε, ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ θα ψηφίσουμε. Και για να είμαι σαφής, ναι σημαίνει αναβολή, όχι σημαίνει να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Right, one ένας ακόμα, μία ψήφος. Πέρα της ψηφοφορίας, έληξε, έληξε η ψηφοφορία. 14 είναι υπέρ της αναβολής, 27 κατά της αναβολής, άρα συνεχίζουμε με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν την έκθεση Tyson. Και μία ακόμα ανακοίνωση έχω. Η συμφωνία για τους, ε, τις συμβιβαστικέ έλεγε ότι θα ψηφίσουμε μόνο τις συμβιβαστικέ και όλες τις άλλες τροπολογίες δεν θα ψηφιστούν. Επί τη βάση αυτής της συμφωνίας λοιπόν πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να επιτρέψουμε προφορικές τροπολογίες που υποβλήθηκαν αργά και να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτές τις τροπολογίες έναντι των τροπολογιών οι οποίες υποβλήθηκαν γραπτός εντός της προθεσμίας. Εάν λοιπόν η προφορική προθεσμία δεν αποτελεί μέρος του τακτικού πακέτου δεν θα τις επιτρέψουμε. Λυπάμαι γι' αυτό αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό, είναι αθέμητο και αντιδημοκρατικό να αφήσουμε να ε, ψηφιστούμε πολύ καθυστερημένε ε, προφορικέ τροπολογίε. όταν έχουμε τι άλλε που υποβλήθηκαν εντό τη προθεσμίας. Ωραία. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση θα αποτανθώ στον εισηγητή και θα ρωτήσω Α, η Μαριάννη είναι εδώ. Θα ρωτήσω εάν είναι μέρος ή όχι του πακέτου η προφορική τροπολογία. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ε, τροπολογία 60. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολο... Ε, συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική γ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Σελίδα 12, συμβαστική ε. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μία διευκρίνηση για αυτή την προφορική τροπολογία του κυρίου Τζιάννη Πιτσέλα. Μαριάν, είναι μέρος του πακέτου αυτό ή δεν είναι. Ή. Αυτή η τροπολογία έχει συμφωνηθεί από τον εισηγητή και τους Σκιώδης. Ένα λεπτό. Α, υπάρχει και δεύτερη του Πιτσέλα. Ε, είναι και αυτή η μέρος του πακέτου τροπολογιών. Μαριάν, για φώτισε μας. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν, λέει η Μαριάν. Τελευταία στιγμή έφτασε σε εμά. Άρα αποσύρεται. Αυτή αποσύρεται. Η πρώτη του πιτέλα είναι στο τραπέζι ή όχι. Ωραία. Η πρώτη τροπολογία λοιπόν ακόμα είναι στο κατάλογο. Η δεύτερη έχει αποσυρθεί. Συγγνώμη, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά Τώρα είναι σαφή διότι ψηφίζουμε την πρώτη προφορική τριπολογία η οποία αποτελεί μέρος του πακέτου. Η δεύτερη αποσύρθηκε. Η πρώτη αναφέρει τις λέξεις εξασφαλίζοντας πάντοτε την ε, προληπτική συνέπεια με το SSM. Αυτές τις λέξεις, ε, αυτή τη διατύπωση προσθέτει. Ωραία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Με την προφορική τοπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ωραία. Προχωρούμε στο τρίτο με τμήμα. Υπέρ. Ο εισηγητής είναι κατά. Άποχες και έγινε δεκτή, έγινε δεκτό το τρίτο, τέταρτο τμήμα υπέρ. Με παρακολουθείτε, είμαστε στο τέταρτο τμήμα. Τέταρτο μέρος τέλος πάντων. Μαριάν, τι γίνεται, είναι στον κατάλογο του εισηγητή. Μείον την προφορική τροπολογία, αλλά υπέρ του τέταρτου τμήματος, που είναι του εισηγητή. Υπέρ, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψηφίζουμε λοιπόν. Όσοι έχουν ένα πλήν, στη λίστα του εισηγητή αυτό ανταποκρίνεται στην προφορική τροπολογία που δεν υπάρχει. Λοιπόν, το τέταρτο τμήμα έχει συν. Άρα ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, έγινε δεκτό. Το τέταρτο μέρος τμήμα. Και το πέμπτο τώρα, το πέμπτο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό και αυτό. Συμβιβαστική Ε, να διευκρινίσω ε, ότι μπορώ να διαβάσω τον κατάλογο ψηφοφορία, αλλά στη δική μου, στο δικό μου κατάλογο δεν υπάρχουν πέντε τμήματα. Τι, ψηφίζουμε, εν πάση περιπτώσει. Ψάχνουμε, ψάχνουμε, αλλά δεν βρίσκουμε. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Μα, θα ήθελα να ξέρω ότι εγώ έχω έναν κατάλογο και δεν τον έχουν οι άλλοι. Να με ενημερώνουν. Από ό,τι φαίνεται. Πιστεύω ότι όλοι Ξέρετε ότι αυτή η συμβιβαστική έχει χωριστεί σε πέντε ε, τμήματα, τα οποία όλα ψηφίστηκαν και όλα έγιναν δεκτά. Μαριάν, κοιτάξτε κυρία Πρόεδρε, στο κατάλογο ψηφοφορία σε αυτό το άρθρο είχε διαιρεθεί σε πέντε τμήματα λόγω των τροπολογιών. Ε, δεχτήκαμε μία προφορική τροπολογία μέρος του πακέτου, η άλλη αποσύρθηκε από τους σοσιαλιστές τώρα, που, τώρα, τώρα στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας που σημαίνει ότι τελικά αυτός ο διαχωρισμός σε πέντε τμήματα δεν χρειαζόταν. Αλλά τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θέλω να ρωτήσω, λέει ο κύριο Λάμπερτ, ότι εσεί ζητήσατε ψηφοφορία ανατμήμα 1, 2, 3, 4, 5. Εμεί ψηφίσαμε πέντε φορέ και δεν ξέραμε περί τίνο πρόκειται, δεν ξέραμε τι ψηφίσαμε. Έλαβα ένα email τώρα στο παραπέντε. Η πρόεδρος. Κανένας δεν μου είπε ότι έχετε, έχω εγώ κάτι στα χέρια μου που δεν έχετε εσείς. Λοιπόν, Ας δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουμε τη συμβιβαστική F με μία αποδεκτή τροπολογία. Δεν υπάρχει ανάγκη διαχωρισμού σε τμήματα. Επειδή αποσύρθηκε η δεύτερη προφορική, ας ψηφίσουμε τώρα όλη την τροπολογία F μαζί με τις λέξεις ενώ ε, θα διασφαλίζει πάντοτε την προληπτική εποπτεία σύμφωνα με τις γραμμές του SSM. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή η συμβιβαστική αυτή. Α, η ε ήτανε. Ε. Τώρα προχωράμε στην F. F. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. το συμβιβαστική G, υπέρ κατά αποχές, δεκτή, H, υπέρ κατά αποχές, δεκτή, συμβιβαστική I, Ι, Υπέρ κατά αποχές δεκτή, Συμβαστική J, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική K, K, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική λάμδα L, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική M, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική N, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ο, όμικρον υπέρ κατά δεκτή. Συμβαστική π υπέρ κατά δεκτή. Συμβαστική Q υπέρ κατά δεκτή. Συμβαστική Ρ R υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική S υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική α, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική ΤΑΦ, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική U και έχω αυτή τη συμβιβαστική U σε έξι τμήματα. Εσείς τι έχετε. Μαριάν. Πρόεδρε, πάλι έχει διαχωριστεί, διότι υπάρχει μια προφορική τροπολογία η οποία δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας των, εισηγητών, των σκιωδών εισηγητών. Άρα μπορούμε να την ψηφίσουμε ολόκληρη και όχι διαχωρισμένη. Η Πρόεδρος, Εντάξει, καλές είναι οι προφορικές τροπολογίες, αλλά δεν επιτρέπουν ε, προφορικές τροπολογίες τη τελευταία στιγμής. Λοιπόν, ε, ο, ο ψηφίζουμε ολόκληρο της τη συμβαστική U, ε, από, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική V. Κάπου, κάπου είναι μέσα στο κείμενο. Ωραία στη δική μου, στο δικό μου αντίγραφο είναι στη σελίδα 40. Συμβαστική V, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική Χ, ε, W, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική Χ, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική Y, Y, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική Z, Z, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα προχωράμε. Συμβαστική ΑΑ και ΑΒ συνδυασμένες είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές. Προχωρούμε στις αιτιολογικές... Α, ε, τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά απορρίπτεται. 61-62. Α, ψηφίζουμε, ψηφίζονται μόνο εάν ε, έχουν περάσει οι 63-64. Λέει. Καταπίπτουν τώρα, τι γίνεται, και 62. Τέλος πάντων, ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 61-62. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AC υπέρ κατά αποχές δεκτή. AD υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική AE αε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ΑΦ ε, δεκτή. AG υπέρ κατά αποχές δεκτή. AH υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική AI υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική AJ υπέρ κατά αποχές δεκτή. AK υπέρ κατά αποχές δεκτή. AL υπέρ κατά αποχές δεκτή. AM υπέρ κατά αποχές δεκτή. AN υπέρ κατά αποχές δεκτή. AO υπέρ κατά αποχές δεκτή. AP υπέρ κατά αποχές δεκτή. AQ υπέρ κατά αποχές δεκτή. AR υπέρ κατά αποχές δεκτή. AS υπέρ κατά αποχές AT υπέρ κατά αποχές δεκτή. AU υπέρ κατά αποχές δεκτή. AV υπέρ κατά αποχές δεκτή. AW υπέρ κατά αποχές δεκτή. AX υπέρ κατά αποχές δεκτή. Y, υπέρ κατά αποχές δεκτή. AZ υπέρ κατά αποχές δεκτή. BA, ε, β' α, υπέρ, κατά, αποχές, BB δεκτή, δεκτή. BC, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προφορική τροπολογία του εισηγητή, που είναι μέρος του, της συμβιβαστικής. 23α, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική BD. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική BE. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. BF. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. BG. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. BH. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. BI υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία του εισηγητή μέρος του συμβαστικού πακέτου, λοιπόν 28α υπέρ κατά αποχές δεκτή. B, G, υπέρ κατά αποχές δεκτή. <coughs> Συμβαστική B, K υπέρ κατά αποχές δεκτή. B.L. L υπέρ κατά αποχές δεκτή. BM υπέρ κατά αποχές δεκτή. BN υπέρ κατά αποχές δεκτή. BO υπέρ κατά αποχές δεκτή. BP υπέρ κατά αποχές δεκτή. BQ υπέρ κατά αποχές δεκτή. BR υπέρ κατά αποχές δεκτή. BS υπέρ κατά αποχές δεκτή. BT υπέρ κατά αποχές δεκτή. BU υπέρ κατά αποχές δεκτή. BV υπέρ κατά αποχές δεκτή. BW υπέρ κατά αποχές δεκτή. BX υπέρ κατά αποχές δεκτή. BY υπέρ κατά αποχές δεκτή. BZ υπέρ κατά αποχές δεκτή. CA υπέρ κατά αποχές δεκτή. CB υπέρ κατά αποχές δεκτή. CC υπέρ κατά αποχές δεκτή. CD υπέρ κατά αποχές δεκτή. CE υπέρ κατά αποχές δεκτή. CF υπέρ κατά αποχές δεκτή. CG υπέρ κατά αποχές δεκτή. CH υπέρ κατά αποχές δεκτή. CI υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το τροποποιημένο κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 47 ψήφισαν, 32 υπέρ, 11 κατά, 4 αποχές. Τώρα θα ψηφίσουμε ε, της ε, τα αιτιολογικά της, του νομοθετικού ψηφίσματος υπέρ, κατά, τι, τι, τι, τι έγινε. Δεν νομίζω ότι αυτό χρειάζεται να γίνει ηλεκτρονικά. Είναι οι αιτιολογικές στην τροπολογία 55. Λομοθετικό ψήφισμα. Τα citations είναι. Λοιπόν, ε, το 55 απορρίφθηκε, το 56 απορρίφθηκε, το 57 απορρίφθηκε, 58 υπέρ κατά απορρίπτεται, 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και τώρα ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τρεις ακόμα, περιμένουμε, τρεις ακόμα πρέπει να ψηφίσουν. Ένας ακόμα. Πέρασε της φοφορίες. 46 ψήφισαν. 31 υπέρ, 11 κατά με 4 αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καθώς αυτό είναι ένα πακέτο μετά από την πρώτη ανάγνωση θα το δούμε και σε σχέση με την έκθεση Γκίγκορτ από κοινού. Λοιπόν. Μπορείτε να χειροκροτήσετε. Πολύ καλή δουλειά έγινε. Ευχαριστούμε. Okay. We will now... Εντάξει και τώρα θα προχωρήσουμε στη συνέχεια με την έκθεση Gigot που θα ψηφίσουμε. Τροπολογίες ε, για τον κανονισμό EBA. Πρέπει να συνεχίσουμε ησυχία παρακαλώ. Συμβιβασμός α, υπέρ. Μια στιγμή. Κατά αποχές εγκρίθηκε ο συμβιβασμός α. Συμβιβασμός β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία Σ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική δέτα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. F υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός I υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μια στιγμή. Τι θα γίνει με αυτά στη μέση. Δεν με σταματήσατε πιο πριν. Λυπούμε. Ας επανέλθουμε. Ας πάμε πίσω στην τροπολογία 187. Τροπολογία 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε θα πάμε στο συμβιβασμό Α, ενώ το κάναμε πριν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμό J, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 204, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός K, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Lα ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός M. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός N Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. εν, 1α. A. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στον συμβιβασμό O. Συμβασμός O υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός O α ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός π υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Q υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 232 υπέρ. Τροπολογία 232 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός R υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός S υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Εντάξει, έχουμε μια τροπολογία προφορική για την 265 τμήμα μέρος του συμβιβασμού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. SB υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 75 και 76 αποσύρθηκαν αυτές οι δύο τροπολογίες. Πάμε τώρα στο συμβιβασμό τι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 270 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 269 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός U υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, να, να το ξανακάνουμε. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 83 και 84 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Όχι, λάθος μου, λάθος μου. 83 και 85 ήταν από κοινού να ψηφιστούν. 83 και 85 που ψηφίσαμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκαν. Και 84 τώρα υπέρ, κατά, όχι καταπίπτει 84, έτσι ή όχι. Ωραία, κατέπεσε η 84, πολύ ωραία. Η ΑΦΚΟ, το της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων, Κατέπεσε και αυτή, τι λέτε. Όχι, οι 83 και 85 εγκρίθηκαν, εντάξει. Ε, τότε πρέπει να την ψηφίσουμε αυτήν, εντάξει. Ωραία. Βιαστήκατε και πήγατε μία παρακάτω. 84, 84 λοιπόν. Α, σωστό. Λέει τα υπόλοιπε, οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Αν οι 83 και οι 85 ε, εγκριθούν, οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Έτσι λοιπόν καταπίπτει η 84 και η, της συνταγματικών υποθέσεων αύκο 1 τροπολογία και αυτή καταπίπτει. Πολύ ωραία. Πάμε στην 86 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 88 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Τοπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 91 και άλλες ταυτόσιμες όχι, 91 και άλλε ταυτόσημες υπέρ. Ναι, 91, 92, έτσι 96. Όλες, όλοι όσοι είναι υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Θα ελέγξουμε, ωραία. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Επειδή πολλοί σηκώνουν το χέρι, το κατεβάζουν, αμφίσιμη η στάση τους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κάποιοι άλλαξαν στάση νομίζω κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας σε πάση περιπτώσει. Λίγη τώρα η ψηφοφορία, εντάξει, απορρίφθηκε, είναι σαφές πλέον τώρα. Απορρίφθηκαν. Ωραία. Πάμε στην 89 ε, τώρα. Έτσι, 89 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε. 90 γι' αυτό ήθελα μόνο σύντομα να πω κάτι. Ο πίνακα για την ψηφοφορία του ΕΛΚ στην 95 και στην 1 έχουμε συν. Πρέπει να μετατραπεί σε πρόσημο πλην, να καταψηφιστούν. Αυτή είναι η σύσταση του ΕΛΚ. Εντάξει, ευχαριστώ. Right. Πολύ καλά λέει η πρόεδρος. Δεν υπάρχει πλέον σύγχυση. 95 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 1. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 90. Τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Αύκο 2. Συγγνώμη, καταπίπτει αυτή, έτσι. Ναι, ναι, λάθος μου. Αύκο 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Εντάξει. Πάμε πάλι πίσω. Λοιπόν, τίποτα δεν κατέπεσε. Για τίποτα δεν έγινε δεκτό, λέει η πρόεδρος. Okay, let's go Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε την 90 λοιπόν. Όλοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Εγώ είχα πει εγκρίθηκε. Μετά είπατε όχι, δεν εγκρίθηκε λέει. Εν, πάση περιπτώσει εγκρίθηκε η 90 κατά πίπτη των συνταγματικών υποθέσεων ΑΦΚΟ 2. 99 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Δεν χρειάζεται γιατί σε σχέση με την 93 που απορρίφθηκε, λοιπόν, δεν χρειαζόταν. Η 98 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Αύκο 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η Αύκο 3. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν σε σχέση με την, αυτή την αιτιολογική σκέψη. Μέχρι, μέχρι πια, μέχρι την 100, 109, έτσι. Ψηφίζουμε την 109 τώρα, τροπολογία. 109. Όσοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Πάμε τώρα στην τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τώρα τροπολογία 107. Υπέρ. 107. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 113 καταπίπτει σε περίπτωση που διαρωτηθήκατε 110 και 111 και αύκο 5 που είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 106 τροπολογία υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ την 106. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορία Αν ψηφίσατε όλοι εντάξει. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 23 υπέρ 18 εναντίον. 112 τροπολογία υπέρ. 112 υπέρ. Κατά. Απόχες. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε λοιπόν. 24 υπέρ 19 εναντίον. Εγκρίθηκε η 112. Αύκο 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Οι υπόλοιπε του εδαφίου 5 της ιτρογικής σκέψης καταπίπτουν. Πάμε στην 122 και 123 υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Πάμε στην 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Εντάξει. 7α. Τώρα η τροπολογία 137 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Η 6 αποσύρθηκε. 128 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Η 132 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 136 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν εκτός από την 135. 135 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Επίσης 130, καταπίπτει 130 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε η 130. 138 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Οι υπόλοιπε σε σχέση με αυτό το εδάφιο καταπίπτουν 8α τώρα, τροπολογία 143 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 144 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Οι υπόλοιπε αυτού του εδαφίου καταπίπτουν. Περνάμε στην 149 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 151 και 152 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 150 πίπτη 153 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή Επιτροπής Προϋπολογισμών G4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τοπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε οι 156 και 158 καταπίπτουν 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 155 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 11 αποσύρθηκε η 11 οι άλλες δύο 159 καταπίπτει 161 δεν καταπίπτει 161 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 162 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Και τώρα θα ψηφίσουμε στο κείμενο όπως έχει τροπολογηθεί. Ηλεκτρονικά η ψηφοφορία άρχεται. 2,1 παραπάνω να ψηφίσει. Λίγη τώρα η ψηφοφορία, κλείνει. Έκλεισε η ψηφοφορία. Συμμετείχαν 43-33 υπέρ, 7 εναντίον, 3 αποχές. Έχουμε κάποια πράγματα που πρέπει να ψηφίσουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Budget 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Budget 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Budget 3 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Όπως το τροποποιήσαμε. Δύο ακόμα να ψηφίσουν. Παρακαλώ ένας ακόμα. Και κλείνει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 34 υπέρ, 7 εναντίον και δύο αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν. Έβγε. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Μαριάν πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να διευκρινίσω μόνο κάτι. Με μεγάλη πλειοψηφία, όπως είδαμε, υιοθετήθηκε η έκθεση για την οποία ήμουν εισηγήτρια και το ίδιο έγινε επίσης και με την έκθεση του Sven Γκίγκολτ, τον οποίο το συγχαίρω φυσικά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι προσπαθούμε από κοινού να βελτιώσουμε την εποπτεία των τραπεζών στην Ευρώπη και να δώσουμε ε, την δυνατότητα η εποπτεία αυτή να αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση τη στιγμή κατά την οποία οι τράπεζες ε, χρειάζονται για να σωθούν τα χρήματα τα κοινοτικά. Προσπαθούμε λοιπόν να καταστήσουμε αποτελεσματική αυτή τη μορφή εποπτείας, αυτός ήταν βασικός στόχος και των δύο εκθέσεων τα κράτη-μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ θα πρέπει να συμμετέχουν στον μέγιστο βαθμό στις διαδικασίες αυτή και στα πλαίσια της συνθήκης και στα όρια της συνθήκης να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Αυτή τη μάχη θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε και στο Συμβούλιο, πιεζόμεθα πλέον χρονικά, Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πετύχαμε τον στόχο μας σε αυτή τη φάση. Αν υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη φάση ή από εδώ και πέρα δεν θα είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς θελήσαμε να προχωρήσουμε πριν το τέλος του χρόνου, συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι είχε πει και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο μπορεί να δουλέψει καλά και γρήγορα, δεν είναι πάντα πολύ εύκολο, μερικές φορές τα πράγματα πηγαίνουν ε, άσχημα ανάμεσα στους κοιόδης εισηγητές, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν ε, επικοδομητικός ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκαν οι σκιώδεις. Φυσικά και αποκλίναμε από τις αρχικές μας θέσεις σημαίνει και ιδέα, αλλά είναι σημαντικό το θέμα και χάρη σε αυτή την εξαιρετική συνεργασία, σαν εισηγήτρια κατέθεσα μια καλή νομίζω έκθεση. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα επιτρέψει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον πιστοτικό κόσμο, προς τον πιστοτικό κόσμο. Κάτι το οποίο το είχε ανάγκη. Σβέν. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν μέρος, ιδιαίτερα στις προσπάθειες της προηγούμενης εβδομάδας. Φυσικά ευχαριστώ την Τάισεν, αλλά και όλους τους κοιόδης. Νομίζω ότι πετύχαμε μια μεγάλη πλειοψηφία, μεγάλη αν λάβει κανείς πόσο ε, αμφισβητούμενο ήταν το θέμα αυτό και αυτό φάνηκε και τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω όμως ότι δεν θα πρέπει να υποτιμάμε την ικανότητα του Κοινοβουλίου να καταλήγει σε συμφωνία για ένα θέμα το οποίο θα παίξει ένα κρίσιμο ρόλο για την έξοδο από την ευρωκρίση και δείχνει και το μέγεθος της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε πλέον να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο επί τη βάση συγκεκριμένων βελτιωτικών προτάσεων δικών μας και όχι μόνο να παραμείνουμε αποκλειστικά στο πλαίσιο των προτάσεων του Συμβουλίου. Αυτό θα αλλάξει λοιπόν τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και αυτό δείχνει ότι η δημοκρατία ανακτάται και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει οικονομική κρίση. Νομίζω ότι αυτό που πετύχαμε μας επιτρέψει να έχουμε κάποιο έλεγχο πάνω σε ένα πακέτο το οποίο στέλνει κάποια ξεκάθαρα μηνύματα μηνύματα τα οποία λέγουν ότι θα υπάρξει στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες εντός και εκτός ζώνης ευρώ και για τον τομέα της Πιστοτικής Ένωσης, της Τραπεζικής Ένωσης. Πιέζουμε για την, θα έλεγα, αποτελεσματική λειτουργία της εποπτικής αρχής των τραπεζών και ταυτόχρονα θα έλεγα υπογραμμίζουμε τις δημοκρατικές ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνει η νέα εποπτική αρχή, παράδειγμα οι ερευνητικές δυνατότητες τις οποίες αποκτά. Καθιερώνεται επίσης και το δικαίωμα έκφρασης των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν αυτή τραπεζική αρχή ε, λειτουργεί επί τη βάση συγκεκριμένων κανόνων σαφώς καθορισμένων. Το πακέτο αυτό προσφέρει αρκετές ιδέες και στο Συμβούλιο και θα προσφέρει στη σταθεροποίηση του ευρώ και της ευρωζώνης. Νομίζω ότι είναι σαφής η εντολή για την διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Δεν θα αποκλείσουμε κανέναν κατά τη διάρκεια αυτής της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν ήταν εύκολη η διαδικασία μέχρι τώρα, αλλά απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Θα πρέπει να γνωρίζει το Συμβούλιο ότι η Συμφωνία για την Πιστοτική Αρχή ε, ε, οφείλεται και στις δικές μας εκθέσεις. Πρέπει να υπάρξει όμως δημοκρατία και από τις δύο πλευρές, πρέπει να το γνωρίζει το Συμβούλιο, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να καταλήξει στις 4 Δεκεμβρίου σε μια κοινή συμφωνία. Η Μάριαν κάτι θέλει να συμπληρώσει. Να επιβεβαιώσω την δική μου θέση ότι και εγώ θέλω μια ξεκάθαρη εντολή για τον τριμερή διάλογο, για την περαιτέρω διαπραγμάτευση να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε γιατί και εσείς είχατε αναλάβει την πρωτοβουλία στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας να υπάρξει ένα πακέτο ε, που αποτελείται από τις δύο προτάσεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά από κοινού. Έχουν συμφωνήσει και τα υπόλοιπα όργανα με αυτή τη λογική. Αυτό έχει σημασία για τη δημοκρατία. Πράγματι επιβεβαιώνω και εγώ ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ήταν ενιαίο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανεξάρτητα από το αν πιστεύουμε και πολλοί από εμά δεν πιστεύουν ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι επαρκή ε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να επιτύχουμε για να προβάλλουμε τη θέση μας. Η απόφαση είναι σαφέστατη, είναι σαφές το τι προκύπτει από την Επιτροπή μας και και οι δύο έχουν δίκιο ε, λέγοντας ότι εδώ πρέπει να κερδίσουμε ξανά την ευρωπαϊκή κουλτούρα, την δημοκρατική διάσταση, τη δημοκρατική διάσταση. Ε, το κοινοβούλιο πρέπει να, να ακουστεί. Η φωνή του κοινοβουλίου πρέπει να ακουστεί. Όταν υπάρχει ένας φάκελος που ανήκει στην ολομέλεια του σώματος για να εκφράσει την φωνή του από κοινού του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, τότε δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από αυτό το ντοσιέ εδώ. Δεν θα υποβάλω αυτή την πρόταση και δεν θα ψηφίσω μια τέτοια πρόταση, διότι η δημοκρατική επιταγή είναι ότι πρέπει να δράσουμε σήμερα, χρειάζονται πράξεις. Όμως είναι απαράδεκτο να ε, αγόμαστε και να από το Συμβούλιο, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρουμε πότε συμβαίνει αυτό και ξέρουμε ποιες είναι οι δυνάμεις πίσω από αυτή την πίεση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρούμε ένα τρόπο απόκρουσης αυτής της πίεσης ή έναν καλύτερο τρόπο να πηγαίνουν τα θέματα στο, στην Ολομέλεια. Πρέπει στο μέλλον να βρούμε μια καλύτερη διαδικασία, μια επίσημη, μια τυπική διαδικασία για να αντισταθούμε ε, σε αυτά τα οποία μας ε, τραβάμε. Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά πρέπει στο μέλλον να γίνει, γιατί τώρα χρειαζόμαστε δράση. Η Πρόεδρος, ήλπιζα ε, ότι θα προχωρήσουμε με την ανάληψη της εντολής δεν πίστευα ότι όλοι σας θέλουν να μιλήσουν. Ήδη μίλησε ένα συνάδελφος από τη σοσιαλιστική ομάδα. Τώρα βλέπω ότι κι άλλοι σηκώναν το χέρι τους. Εκτός αν υπάρχει διαδικαστικό θέμα, δεν θέλω να ε, μιλήσουν όλοι, να δώσω αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, συμφωνείτε με συνένεση όλοι να προχωρήσουμε στον τριμερή διάλογο με την ε, συνήθη ομάδα, εισηγητής, σκιώδης εισηγητής. Συμφωνούμε λοιπόν, υπάρχει συνένεση υπ' αυτού. Ε, αντιρρήσεις, εγώ έχω μία αντίρρηση, βλέπω, και ε, θα την ψηφίσουμε. Θετική ψήφο σημαίνει ότι προχωρούμε με την εντολή, τη διαπραγματευτική εντολή για την πρώτη ανάγνωση. Ψηφίζουμε αυτό. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε την εντολή για τη διαπραγματευτική εντολή. Ναι σημαίνει ναι στη διαπραγμάτευση πρώτη ανάγνωση. Όχι σημαίνει ότι θέλετε να πάει στην Ολομέλεια. Ε, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 33 υπέρ, μία ψήφος κατά, πέντε εποχές. Ωραία. Συμφωνούμε για την πρώτη ανάγνωση. Ε, θα γίνει λοιπόν ε, η διαπραγμάτευση συμφωνίας για την πρώτη ανάγνωση. Την πρώτη ανάγνωση. Επίσης θέλω να πω εκ μέρους του Προεδρείου ότι ό,τι καταφέραμε το καταφέραμε μέσα σε ένα πολύ πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα Είχαμε πολλές συνεδριάσεις που κράτησαν μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέρα με τη μέρα ε, εργαστήκαμε σκληρά και τώρα αναμένουμε μία, ε, ένα πλήρες ολοκληρωμένο μια πλήρη ε, διαπραγματευτική εντολή ε, το Δεκέμβριο για να αρχίσουμε τον τριμερή διάλογο. Δεν ε, αναμένω έναν μερικό, έναν, μια μερική εντολή, μια ολοκληρωμένη 100% διαπραγματευτική εντολή για τον Δεκέμβριο. Το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αποτελεί μέρος της, κανείς, της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Εμείς ακολουθούμε τη διαδικασία που επιβάλλεται από τις συνθήκες. Εμείς διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο. Εάν δεν το επιτύχουμε τότε θα υπάρχει ευθύνη στους ώμους του Συμβουλίου ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ότι δεν θα επιτύχουμε να τηρήσουμε την προθεσμία του Δεκεμβρίου. Η Μαριάννα. Ε, κυρία Πρόεδρε, ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα για το οποίο εργαστήκαμε τόσο σκληρά. Πριν όμως ε, συνεχίσουμε με την επόμενη ψηφοφορία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τα μέλη της γραμματείας διότι εργάστηκαν πραγματικά πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρουμε ό,τι καταφέραμε. Και χτες και κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας ήταν εξαιρετικά ε, πρόθυμοι να βοηθήσουν, εξαιρετικά εργατικοί και ευχαριστώ πάρα πολύ τη γραμματεία και όλα τα στελέχη αυτού του σώματος. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα προχωρούμε σε έναν άλλο σημαντικό φάκελο, την τελευταία ψηφοφορία. Η έκθεση της κυρίας κυρίας Γκουλάρ. Θέλετε το λόγο. Λίγα λόγια, αν είναι δυνατόν. να εξηγήσω εν πάση περιπτώσει γιατί υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής. Συνεργαστήκαμε στενά τις τελευταίες εβδομάδες με τους Κιώδης, τους οποίους ευχαριστώ. Την τελευταία στιγμή όμως κατετέθησαν ε, αιτήματα από πλευρά των ΣΕΡΠΑ. Ε, δεν προβλέπεται από τον κανονισμό, αλλά στα πλαίσια ενός επικοδομητικού πνεύματος προσπαθήσαμε να τις εντάξουμε στο κείμενο. Εγώ ήμουν ανέκαθεν δεκτική αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές να είναι πραγματικά οι συνομιλητές της κάθε πολιτικής ομάδας επί του προκειμένου κειμένου. Δέχτηκα, όπως είπα, στα πλαίσια ενός συμβιβαστικού πνεύματος να λάβω υπόψη αυτά τα οποία μου ζητήθηκαν. Αλλά για να δουλεύουμε σωστά από εδώ και πέρα θα πρέπει να, ε, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τους σκιώδεις και τους συνεισηγητές. Όπως είπε και η Μάριαν, η διαδικασία έχει επιβαρύνει και τη γραμματεία και τους συνεργάτες. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους λοιπόν, γιατί ανεξαρτήτως της επιθυμίας του εισηγητή και των σκιωδών αναγκάστηκαν την τελευταία στιγμή πολύ βιαστικά να κάνουν πράγματα. Εν δεν το κάνουμε θέμα, θα προχωρήσουμε με πνεύμα συμβιβασμού. Αλλά πρέπει να το ε, συγκεκριμενοποιήσω το θέμα όλα θα πρέπει να ακολουθούν μία τάξη, να σέβονται μία τάξη. Okay, there are one or two, uh, Καλώς. Πράγματι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία όταν φτάσω θα πρέπει να σταθούμε λίγο και αναφέρεται ακριβώς στη συμφωνία των Σέρπα στην οποία αναφέρθηκε η ε, Σιλβί. Σιλβή. Καλώς. Λοιπόν ξεκινάμε παρακαλώ. Καταρχάς, προφορική τροπολογία στη συμβιβαστική Α από τους σοσιαλιστές. Μπορεί παρακαλώ να γίνει δεκτή η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συμβιβαστική Α. Τι είναι υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε το σύνολο της συμβιβαστικής... Θέλεις να ψηφίσουμε ξεχωριστά την προφορική τροπολογία. Η κυρία Γκουλάρ θέλει να ψηφιστεί ξεχωριστά λοιπόν η προφορική. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η προφορική. Συνεχίζουμε λοιπόν με την A. Χωρίς την προφορική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική C. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. D υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ή e, αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία στην F. Λοιπόν, ξεχωριστά. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική F, αγγλικό, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική G, αγγλικό, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική H, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 80. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές δεκτή. J υπέρ κατά αποχές δεκτή. K υπέρ κατά αποχές δεκτή. L αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα στην παράγραφο 6 υπάρχει μια προφορική τροπολογία στην συμβιβαστική M ε, για να υπάρχει σύμπτωση με την έκθεση των Σέρπα και Βαν Θα σας διαβάσω το νέο κείμενο. Υπογραμμίζουμε ότι όλες, όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά μέσα, οι θεσμοί, τα οποία σένστο στρίκτο ή σένσο λάτο αποτελούν τμήμα του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, θα πρέπει να νομιμοποιηθούν με δημοκρατικό τρόπο Λοιπόν, αυτή είναι η προτινόμενη προφορική τροπολογία. Εάν γίνει δεκτή, θα αντικαταστήσει ουσιαστικά την συμβιβαστική πρόταση M αγγλικό. Θέλετε να σας ξαναδιαβάσω ή ακούσατε αυτό που είπα. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 98. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 100 αν και είμαι βέβαια ότι απερίφθη. Πέρα της ψηφοφορίας για την 100. 17 υπέρ 23 κατά. Πράγματι απερίφθη. Συμβιβαστική εν αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΥΜΚΟ 14 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 116 αν και νομίζω ότι γίνεται δεκτή. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκαοκτώ υπέρ, 20 κατά απερίφθη. 117. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 117 η οποία βέβαια νομίζω ότι απορρίπτεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 14 υπέρ 26 κατά. Απερίφθη. Συμβιβαστική ο αγγλικό σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής τροπολογίας ΟΟΥ Αγγλικό. Ψηφίσατε όλοι. 18 υπέρ 22 κατά. Το δεύτερο τμήμα κατέπεσε. Τροπολογία τώρα 120. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α, όχι. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος πάλι για την 120. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 26 υπέρ 14 κατά. 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές δεκτή 128 υπέρ αλλά εδώ έχω την προφορική τροπολογία στην 128. Συμφωνείτε με το, η ψηφοφορία της ε, προφορικής. Καλώς λοιπόν. Ας ψηφίσουμε τώρα την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η, ψηφοφο... η τροπολογία, η προφορική γίνεται δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογημένη τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 129 υπέρ κατά αποχές δεκτή 130 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απερίφθη αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 130 ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας Πράγματι απερίφθη 17 υπέρ 24 κατά. Τροπολογία 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική π υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική Q υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Λοιπόν, στην συμβιβαστική R αγγλικό υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Ας ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν προστίθεται λοιπόν αυτή η προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική R. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή αν και θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 22 υπέρ 19 εναντίον. Συμβιβασμός Α. Πώς είπατε? Συγγνώμη, αυτό μόλις το ψηφίσαμε. Συμβιβασμός S λοιπόν, υπέρ. Κατά. Έχει δημιουργηθεί κάποια σύγχυση. Μπορείτε να επικεντρωθείτε, να προσέξετε και να σηκώνετε τα χέρια έγκαιρα. S υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός T υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 160 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 158 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 161 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε αλλά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας Τρει τώρα που ήταν, τέλο πάντων, απορρίφθηκε. 18 υπέρ, 21 εναντίον. Συμβασμός U υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 170 τοπολογία. Προφορική τροποποίηση αυτής αλλάζει την Ευρωζώνη σε Ευρωομάδα, Eurozone to Eurogroup. Αποσαφήνιση αυτή σχετικά. Ψηφίζουμε την 170 με την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά, αποχές, νομίζω καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αυτό που ψηφίζουμε είναι η τροπολογία 170, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας, αποτέλεσμα, καταπίπτει. Ισοψηφία 21-21. Απορρίπτεται. Πάει αυτή. Εντάξει. Τροπολογία 171 τώρα. Υπέρ. Κατά. Μπορούμε να ελέγξουμε και αυτήν ψηφίζουμε την 171 ηλεκτρονικά άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εντάξει. Απορρίφθηκε. 16 υπέρ, 26 εναντίον. Τροπολογία 172 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα έχουμε μια προφορική τροποποίηση στον συμβιβασμό Β προσθέτει και μηχανισμός ε, καταθέσεων, ευρωπαϊκός μηχανισμός εγγύσεων καταθέσεων. Όλοι λοιπόν όσοι είναι υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε τους αριθμούς τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 25 εναντίον. Απορρίφθηκε λοιπόν. Συμβιβασμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 185 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Την 185. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε λοιπόν 16 υπέρ 25 εναντίον. Τροπολογία 186 υπέρ κατά Μακάρι να έβλεπα περισσότερους να σηκώνει το χέρι τους. 186 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 20 υπέρ 22 εναντίον απορρίφθηκε. 187 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 188 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 190 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 191 για διαγραφή όσοι είναι υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. 20 υπέρ, 21 εναντίον. Απορρίφθηκε λοιπόν. Πού πάμε τώρα. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στην 195 τροπολογία. 195 υπέρ Βρήκατε όλοι, όλοι εντάξει κατά, μετά το υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 196 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Προφορική τροποποίηση λοιπόν για την τροπολογία 197 αξιόπιστα λοιπόν σχέδια για και τα λοιπά. Ψηφίζουμε την προφορική τροποποίηση ξεχωριστά για την προσθήκη αυτών των λέξεων. Όσοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεν θα, προσθεθούν αυτά στη διατύπωση. Καταψηφίστηκε η προφορική τροποποίηση. Τροπολογία 197 ξεχωριστά τώρα, χωρίς τροποποίηση ή προσθήκη. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και άρχεται η ψηφοφορία. 197. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 18 εναντίον. Εγκρίθηκε. Και πάμε τώρα στην 198 τροπολογία. Υπέρ. 198. Εντάξει, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 199 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 200 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός W υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 211 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 213 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 213 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε 15 υπέρ 25 εναντίον. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα πάμε στην προφορική τροποποίηση στο συμβιβασμό Y. Προφορική πρόταση. Λοιπόν, αυτό που βρίσκεται υπογραμμισμένο με παχιά γράμματα στο κείμενο. Λοιπόν, εντάξει, θα σας το διαβάσω για να διευκρινιστεί το σύνολο αυτού που θα ψηφίσουμε τώρα. Αν είμαστε υπέρ, αν είσαστε υπέρ της ε, τροποποίησης, τροπολογίας Y, για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμα μέτρων για να διεξέλθουμε από την κρίση και μεταξύ των πρώτων βημάτων του δεσμευτικού χάρτη πορείας και θα πρέπει η συνέχεια να γίνεται με βάση την κανονική νομοθετική διαδικασία με πλήρη ε, νομοθετική δημοκρατική λογοδοσία σε σχέση με την λήψη απόφασης. Προετοιμάζοντας αυτές τις αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει ένα προσωρινό σώμα που θα συναπατήσει από ευρωβουλευτές, εκπροσώπους των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει πλήρη χρήση των εξουσιών του μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία και του δικαιώματός του να ξεκινήσει να οδηγήσει σε αλλαγές της συνθήκης. Αυτό το σώμα θα εξετάσει και την δυνατότητα διασφάλισης γενικών ομολόγων που θα λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο ενός διευρυμένου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτό θα ψηφίσουμε τώρα ως πρόταση. Και αν είσαστε υπέρ αυτής της πρότασης, τότε η αρχική, τροπο, ε, η αρχική τροπολογία Y θα καταπέσει. Όσοι είναι υπέρ λοιπόν αυτού του κειμένου, κατά αποχές, εγκρίθηκε αυτό το κείμενο. Και το υπόλοιπο του συμβιβασμού Y αντικαθίσταται έτσι. Και περνάμε στην τροπολογία τώρα Συγγνώμη, 224 διορθώνει η πρόεδρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια 225 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά κατά αποχές. Νομίζω εγκρίθηκε, αλλά θα ψηφίσουμε το δεύτερο ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα της 225 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Δεύτερο τμήμα της 225 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Ακαταπίπτει. Ε, απορρίφθηκε για την ισοψηφία 21-21 και πάλι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πολύ καλά. Τροπολογία 226 υπέρ. 226 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 228 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές φαίνεται ότι απορρίφθηκε. Αλλά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε και άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 20-20 πάλι ισοψηφία απορρίφθηκε. Πάει και αυτή. Καταπίπτει λοιπόν. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Της νομικής επιτροπής ε, παράγραφο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε, η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε, ΙΜΚΟ για την, το τρίτο εδάφιο εγκρίθηκε, ΙΜΚΟ εδάφιο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε το εδάφιο 7 της ΣΥΜΚΟ. Κάποιοι δεν σήκωσαν τα χέρια τους επαρκώς. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ακόμα. Συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά. Πέρα ψηφοφορία τώρα απορρίφθηκε λοιπόν. 15 υπέρ, 24 εναντίον. Απορρίφθηκε. Διορθώθηκα λοιπόν. Ευχαριστώ. Παράγραφος 8. Ήμκο υπέρ κατά αποχές, να ελέγξουμε πάλι. Εδάφιο 8 της ΣΥΜΚΟ, δεν σηκώνουν αρκετοί τα χέρια τους. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται, παράγραφος 8. Ψηφίσατε όλοι, ένας ακόμα ακόμα και κλείνουμε την ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα και αποτέλεσμα απορρίφθηκε 19 υπέρ 20 εναντίον. Ήμκο εδάφιο 9 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε και πάλι εδάφιο 9 ΙΜΚΟ ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Τώρα θα κλείσουμε την ψηφοφορία. Δύο που δεν έχουν συμμετάσχει ακόμα. Απορρίφθηκε. 17 υπέρ, 22 εναντίον. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 231 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 232 υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 232. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Μια στιγμή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι. Ψηφίσατε όλοι τώρα. Συνεχίστε να ψηφίζετε. Αρκετοί ακόμα. Τρει, δύο που απομένουν. Κλείνω την ψηφοφορία τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Και απορρίφθηκε. 16 υπέρ, 20 εναντίον. Απορρίφθηκε. Αρχικό κείμενο τώρα σε σχέση με τον τίτλο του παρατήματος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Z σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα <clears throat> του συμβιβασμού Z ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και απορρίφθηκε. 16 υπέρ, 22 εναντίον απορρίφθηκε. Τη τελευταία στιγμή προφορική τροποποίηση. Καλύτερα να σα τη διαβάσω για το παράτημα. Τι λέει. Λέει το 1-2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την άμεση θέσπιση ενός συστήματος για την... με βάση τις εξής αρχές θα προβλέπει τη συμμετοχή ε, ε, μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων, όπως προβλέπεται από τους συνταγματικούς κανονισμούς των εμπλεκομένων κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα, τα οποία θα αναφέρονται στην τελική έκθεση Φαν για μια αυθεντική οικονομική και νομισματική ένωση. Αυτό θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα, αντί του αρχικού κειμένου. Εν περιπτώσει, επ' αυτού θα ψηφίσουμε όσοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεν ξέρω πώς αποκαλείται. Είναι τώρα ένα β ένα 1-2. Παίρνουμε τώρα την προφορική τροποποίηση για τον συμβιβασμό ΑΑ από πλευράς των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Στο δεύτερο, στη δεύτερη παύλα προστίθεται όσον αφορά άμεσα την άμεση συμμετοχή των κρατών μελών. Το πιο εύκολο θα είναι απλά να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ψηφίζουμε ξεχωριστά. Αυτοί που συμφωνούν άμεσα, άμεση συμμετοχή να ενταχθεί. Όσοι είναι υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για να είναι απόλυτα σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονικά. Εντάξει, τέλος ψηφοφορίας τώρα. Απορρίφθηκε. 16 υπέρ, 25 εναντίον. Δεν θα μπει το άμεση ή άμεσα μέσα. Επίσης, θέλω να διαγραφεί η λέξη forfeit fund και θα αναφέρεται επαρκώς θα υφίστανται κυρώσεις. Όσοι είναι λοιπόν σε σχέση με αυτή την πρόταση υπέρ, κατά, αποχές, δεν δεχόμαστε ούτε αυτή την προφορική τροποποίηση. Απορρίφθηκε λοιπόν. Ο συμβιβασμός ΑΑ λοιπόν με, χωρίς τροποποίησης υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ναι, κάπου στη σελίδα 33. Έχουμε το συμβασμό ΑΒ, AB. Όσοι είναι υπέρ αυτού, κατά αποχές εγκρίθηκε. AC υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. AD υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Το 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 14 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε το 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 22 υπέρ 17 εναντίον. Και πάμε τώρα στην τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 17 υπέρ. Κατά. Απόχες. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 17 ηλεκτρονικά. Άρχεται. 17 ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 18 υπέρ, 22 εναντίον. Απορρίφθηκε. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μα επιτέλους πρέπει να ελέγξουμε την 18 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε την 18. Ψηφίσατε όλοι. Ναι, ναι, ψηφίζουμε την 18. Λίγη ψηφοφορία, έληξε η ψηφοφορία, αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 15 υπέρ, 22 εναντίον, απορρίφθηκε. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 20 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεν χρειάζεται το αρχικό κείμενο. Έτσι. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε την 21. Να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τρεις ακόμα που απομένουν. Δύο. Λίγη τώρα η ψηφοφορία. Τελευταία ευκαιρία να πατήσετε το κουμπί. Έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 21 υπέρ 18 εναντίον. Εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε την 22. Δεν συμμετείχαν ξεκάθαρα όσοι σήκωναν τα χέρια. 22 ηλεκτρονικά άρχεται. 22. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 24 υπέρ, 15 εναντίον. Εγκρίθηκε. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 24 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 24 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Δεκτή. 18 υπέρ, 17 εναντίον. Δεκτή. 25 υπέρ. Κατά. Είναι πολύ δύσκολο άμα δεν σηκώνετε ξεκάθαρα τα χέρια. 25 πάλι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 27 υπέρ, κατά 27 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 27 28 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 28 ψηφίζοντας ηλεκτρονικά άρχεται 2,1 που απομένει Λίγη τώρα η ψηφοφορία. Έκλεισε, έληξε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 19 υπέρ, 21 εναντίον. Απορρίφθηκε. 29 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Εντάξει, τώρα πάμε στην τροπολογία 30. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια προφορική τροποποίηση να ενταχθεί η λέξη παγίωση, consolidation. Θα την ψηφίσουμε ξεχωριστά. Όσοι είναι υπέρ του να προσθεθεί το consolidation, υπέρ της προσθήκης, κατά αποχές η προφορική αυτή τροποποίηση εγκρίθηκε. Με την προφορική τροποποίηση τώρα στην τροπολογία 30 ψηφίζουμε την 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε η 30. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίφθηκε αλλά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 31 ηλεκτρονικά. Άρχεται παρακαλώ. Δύο ακόμα που απομένουν. Συνεχίστε. Λίγη ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Ωραία. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. 13 υπέρ 24 εναντίον. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 32 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 32 και άρχεται η ψηφοφορία. Όλο και φθήνει ο αριθμός των συμμετεχόντων και είναι όλο και πιο δύσκολο. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 23 υπέρ, 16 εναντίον. Έτσι λοιπόν πράγματι εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές στεκτή. Προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 2. Η προφορική τροποποίηση θέλει να προσθεθεί το εξή στο κείμενο. Λέει με την εξαπλή πρόταση και την μελλοντική διπλή πρόταση και την κοινοτικοποιημένη συμφωνία για τα δημοσιονομικά σύμφωνα με το άρθρο 16 του TSCG. Μα τι σημαίνει αυτό κοινοτικοποιημένη, διότι δεν είναι αγγλικά αυτό το communitarized, νομίζω σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο σημαίνει αυτό λέγει η πρόεδρος, απλά έτσι. Νομίζω είναι communitized που ήθελα να πούν και όχι communitarized. Νομίζω πρέπει αυτό να χτενιστεί και να σημαίνει όπως εννοεί σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο που θα ακολουθηθεί. Εν πάση περιπτώσει, είτε είσαστε υπέρ είτε κατά. Παίρνουμε λοιπόν πρώτα την προφορική τροποποίηση. Όσοι είναι υπέρ αυτή. Κατά. Άποχες. Θα ελέγξουμε ψηφίζοντας ηλεκτρονικά αυτή την προφορική τροποποίηση. Άρχεται. Άρχεται. Είναι μόνο για την ένταξη, την προσθήκη της προφορικής, του κειμένου της προφορικής τροποποίησης. Τίποτα άλλο. Εντάξει, επ' αυτού μόνο για το αν θα τροποποιηθεί με την προφορική προσθήκη αυτή ή όχι. Λοιπόν, δεν μας αρέσει το Community communitarized, εφόσον δεν είναι αρεστό αυτό, απορρίπτεται. Επανερχόμαστε στην αρχική τροπολογία 2, λοιπόν, ως είναι υπέρ αυτής. Αρχική τροπολογία 2, υπέρ. Έτσι, μια στιγμή. Εντάξει, εναντίον τώρα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2. Λοιπόν, τροπολογία 2, χωρίς προφορική τροποποίηση, υπέρ της 2. Κατά. Άποχες. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 2 και άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Μάλιστα, πολύ καλά. Τώρα, νομίζω θα έλεγα ότι πρέπει να... Όχι, πάμε στον συμβιβασμό AE, όσοι είναι υπέρ. Συμβιβασμός Παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου. Μα το κάναμε το αρχικό κείμενο σε σχέση με την τροπολογία 2. Τελείωσε. Πάει η 2. Λοιπόν, είχε η πρώτη τροπολογία εγκρίθηκε η 1. Το, η 2 εγκρίθηκε. Πάμε στον συμβιβασμό AE. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 3. Όχι. Όχι. Συμβασμός AF. Συμβασμός AF πρώτα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 τώρα. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Κάποιος θέλει να ελέγξουμε την 3. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 3 ηλεκτρονικά και άρχεται. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 3. Δύο ακόμα που απομένων. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί. Τώρα λύγει λίγο η ψηφοφορία και έληξε, εγκρίθηκε, 19 υπέρ 18 εναντίον, εγκρίθηκε. Επειδή κάποιοι δεν πατούν το κουμπί έγκαιρα, υπάρχει αυτή η διαρροή. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Αιτιολογικό 2 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 7 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε τροπολογία 7. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Λυπάμαι πολύ, ζητώ συγγνώμη, είναι πολύ δύσκολο. Δεν σηκώνετε ξεκάθαρα τα χέρια, συζητάτε, δεν μπορώ να δω τι συμβαίνει. Τροπολογία 7. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε 17 υπέρ 21 εναντίον. Πάμε στο αρχικό κείμενο, στο 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, αρχικό κείμενο στο 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, αρχικό κείμενο στο 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα η τελική ψηφοφορία επί του κειμένου όπως το τροποποιήσαμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Ένας ακόμα που απομένει. Συνεχίστε. Τελευταία σας ευκαιρία. Λίγη τώρα η ψηφοφορία όπου να είναι. Ωραία, έληξε. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 19 υπέρ, 12 εναντίον, 7 αποχές. Συγχαρητήρια Σιλβί, σας ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα υπό τα διάφορα και η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 3 Δεκεμβρίου το απόγευμα. 3 με 6.30 και μετά την Πέμπτη 9 με 12.30. η 6 Δεκεμβρίου.